Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με την ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς λοιπόν καλώς ήρθατε στην κοινή συνεδρίαση ΕΚΟΝ Ο κύριος Γουαλτιέρη δεν μπορεί να έρθει σήμερα το πρωί. Βρίσκεται σε μια συνεδρίαση στην Ιταλία. Έχουμε τον αντιπρόεδρο όμως Επιτροπής ΕΚΟΝ μαζί μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην κοινή αυτή συνεδρίαση ΕΚΟΝ και ΛΥΜΠΕ. Όσον αφορά τη σημερινή ψηφοφορία, έχουμε ένα σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με τον άρθρο 153 του κανονισμού σχετικά με τον κατεξοδότηση κανονισμό της Επιτροπής 24 Νοεμβρίου 2016 για τροποποίηση του κατεξοδότηση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016 1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2015 849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες. Ξέρετε ότι η Γουιάννα απομακρύνθηκε από τον τελευταίο αυτό κατάλογο σύμφωνα με το πόρισμα της ομάδας χρηματοπιστωτικής δράσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, το είπαν αυτό και οι συντονιστές όσον αφορά την πρόταση αυτή και υπάρχει η δυνατότητα απόρριψη τη κατεξοδότηση αυτή τη πράξη. Προτού λοιπόν τη σημερινή ψηφοφορία, να σα πω λίγο ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Παράταση τη προθεσμία κοινοβολευτικού ελέγχου έχει ζητηθεί για ένα, μήνα ακόμα, άρα η προθεσμία για την επίσημη απόρριψη τη πράξη αυτή είναι 24 Ιανουαρίου 2017 και το σχέδιο ψηφίσματος που θα ψηφίσουμε σήμερα θα περάσει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου του 2017. Έτσι λοιπόν η ΕΚΟΝ και η ΛΥΜΠΕ υπέβαλαν σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για το οποίο λάβαμε μάλιστα και τροπολογίες. Ας ψηφίσουμε λοιπόν πρώτα τις τροπολογίες και στη συνέχεια το σχέδιο ψηφίσματος. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Ο συμπρόεδρος θέλει να κάνει μια σύντομη ανακοίνωση. Ευχαριστώ κύριε Μωράες. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος του Πρόεδρος της δικής μας Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας στην 1α. Απευθύνομαι στα μέλη της ΕΚΟΝ. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε με την ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Παράγραφος 1, αρχικό κείμενο, άρτη ψηφοφορία. Ηλεκτρονική θα γίνει ψηφοφορία για όλα τα σημεία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα λεπτάκι. Έχουμε και τα μέλη της Επιτροπής ΣΕΚΟΝ. Προτού ξεκινήσουμε, όσοι... Ένα λεπτό, κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ πολύ. Όσοι δεν έχετε την κάρτα ηλεκτρονική ψηφοφορίας μαζί σας, πείτε το μου τώρα σας παρακαλώ. Εσεί έχετε την κάρτα σας μάλιστα. Για τους τρεις λοιπόν συναδέλφου που δεν έχουν μαζί τους την κάρτα τους, σας παρακαλώ πολύ ψηφίστε διανατάσεως εσείς οι τρεις και θα καταγράψουμε την ψήφο σας. Όλοι οι υπόλοιποι είστε εντάξει. Πολύ ωραία. Ψηφίσουμε πάλι την πρώτη παράγραφο Παράγραφος 1. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος πέρθμων 4. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Λειτουργική αναφορά υπαριθμών 1. Αρχικό κείμενο. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά υπαριθμών 2. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά υπαριθμών 3, άρτη ψηφοφορία. Πέρα Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά υπαριθμών 4, άρτη Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 4α νέα, τροπολογία υπαριθμών 1, άρτη ψηφοφορία. Πέρα Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά υπαριθμών 5. Άρτη ψηφοφορία. Πέρα Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 6. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 6α. Νέα τροπολογία υπαριθμών 2. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τελική αναφορά 7α νέα τροπολογία 3 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τελική σκέψη α άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τελική σκέψη α α μικρό, νέα, τροπολογία 4, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΒ, νέα, τροπολογία 5, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ετολογική σκέψη Β, άρθρη ψηφοφορία. Πέρα. συγκρίνεται. σκέψη ΒΑ. Νέα τροπολογία 6. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. σκέψη Σ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ετολική σκέψη ΣΑ νέα τροπολογία 7 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ετολική σκέψη ΣΒ νέα τροπολογία 8 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ετολική σκέψη D άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ετολική σκέψη DA νέα τροπολογία 9 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη E, τροπολογία 10, άρτη ψηφοφορία. Πέρας κρίνεται. Το αρχικό κείμενο τώρα, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Έχετε δίκιο, μπορούμε να αφήσουμε εκτός το αρχικό κείμενο. Περνάμε στην τροπολογία 11, τη λογική σκέψη ή e, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. εταιρεολογική σκέψη F, τροπολογία 12 δηλαδή, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13, άρτη ψηφοφορία. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 13, λέει ο πρόεδρο. Σα ζητώ συγγνώμη. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Άρτη ψηφοφορία. περα Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 τώρα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μονομαστική κλίση τώρα, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ, το σύνολο του τροποποιημένου κειμένου. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 υπέρ, 8 κατά, 25 αποχές. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως σας είπα, το κείμενο αυτό θα περάσει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου του 2017. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΕΚΟΝ για την παρουσία τους και εμείς ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα προχωρήσουμε με την ψηφοφορία άλλων κειμένων. Προετοιμαζόμενοι λοιπόν την ψηφοφορία.